στο διάλογο της με την Ουγγαρία στα θεμελιώδη δικαιώματα. Αν δεν συζητηθεί αυτό το κείμενο, δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα που θα άξιζε να ασχοληθούμε με αυτό για την Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Σημειώνω λοιπόν ότι υπάρχει πρόταση για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Θα παραπευθεί στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, που θα λάβει και τη σχετική απόφαση. Ας περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έκθεση Κορέρα. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. La votazione è chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Άουκεν. Δεν θα γίνει τώρα συζήτηση. Δεν έχει προβλεφθεί συζήτηση στην ημερήσια διάταξη για την Ουγγαρία. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Διαδικαστικό. Παρακαλώ. Please, point of order. Διαδικαστικό. Το Κοινοβούλιο και η Ολομέλεια είναι κυρίαρχη στην αρχή κάθε συνόδου να αποφασίζει για τη διάταξη των εργασιών και τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. La proposta è chiara. Η πρόταση είναι σαφέστατη, αλλά σε αυτή τη φάση ο πρόεδρος είναι αρμόδιος να λάβει απόφαση. Θα παραπέμψω λοιπόν την πρόταση αυτή στον πρόεδρο ο οποίος θα λάβει την απόφαση και θα την κοινοποιήσει στην Ολομέλεια. Η Επίτροπος Ρέντινγκ ζήτησε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, η Ολομέλεια έχει μόλις ψηφίσει μια έκθεση, την έκθεση κουρέα de και θα ήθελα εξ ονόματο της Κομισιόν να κάνω την εξή δήλωση. Καταρχήν η Κομισιόν χαιρετίζει τη συμφωνία που επετέφθη με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και την, ε, όπως προκύπτει από την έγκριση της έκθεσης Korea de Campus και προσβλέπουμε σε μια ταχεία περάτωση των διαδικασιών για αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιλεξιμότητα σχεδίων κοινού συμφέροντο για χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τη διαμεθοριακή υποδομή ενέργεια, η Κομισιόν θέλει να τονίσει ότι θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι εθνικέ αρχέ να καλύπτει και χρηματοδοτήσει σχεδίων κοινή ωφελία που βελτιώνει τη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας και η Κομισιόν επιφυλάσσεται του δικαιώματο να κάνει προτάσει συγκεκριμένε στα θέματα αυτά επί τη βάση της ε, εμπειρία που έχει κτηθεί από την παρακολούθηση των προηγουμένων αυτών θεμάτων και βάσει του άρθρου 16 για τις κατευθυντές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και δομέ ενέργεια. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Περνάμε στην έκθεση Όκεν. Ε, δίνετε να λάβει το λόγο αν το επιθυμεί κυρία Συγγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε δεν είναι τόσο συχνό μία ε, ειδική έκθεση να είναι έκθεση του Κοινοβουλίου και κρίμα που δεν έγινε πλήρη συζήτηση όπως ε, θα έπρεπε. Πρόκειται για ε, το σεβασμό των πολιτών και τη συμμετοχή των πολιτών. Είναι ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και καλό θα ήταν να την ακούγαμε. Καλή είναι η έκθεση που προέκυψε από την Επιτροπή μας. Ε, πρόκειται για ε, δύο ζητήματα. Ε, η Αυστρία ε, έχει δεσμευθεί ε, ε, να ακολουθήσει ε, μια πιο μεγάλη διαδικασία με ειδική ανάλυση εκ των προτέρων για το αεροδρόμιο της Βιέννης. Αφήστε που δεν είναι εκ των προτέρων, είναι εκ των υστέρων για να μην πω και νεκροψία γιατί είναι ήδη πολύ έργα Αλλά οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να προσφεύγουν ε, αρμοδίως εξού ε, και η προσφυγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και θα πρέπει να το τονίσουμε. Ε, χρειάζεται αναθεώρηση της αντίστοιχης οδηγίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πλαίσιο για δράσεις περιβαλλοντικές. θα πρέπει να τηρούνται όλα τα κριτήρια για τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Και πιστεύω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει εμείς να ε, υπερασπιζόμαστε στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Ήταν ε, πολύ μεγάλη πλειοψηφία και βεβαίως ε, καλείται τώρα να διορθώσει ε, αυτές τις στρεβλές καταστάσεις η Ευστρία. Ελπίζω στο μέλλον να προβλέψουμε και κυρώσεις για να μην υπάρχει επανάληψη. Μάλιστα. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Αρσένη. Τροπολογία. Πρώτο μπλοκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροποποιηθήσα πρόταση επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Ε, τελικό. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Credo sia approvata. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται έκθεση Eichhout. Πρώτο μπλοκ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, della... Πρόταση τροποποιηθέσα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρόταση Επιτροπής. Τώρα σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Απροβάτο. Εγκρίνεται. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα και ο κύριος Μπρόκ έχει πρόβλημα με το μηχάνημά του. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ξέχασα την κάρτα ψηφοφορίας. Υπερψήφισα και τις δύο εκθέσεις ονομαστικές και τις επόμενες ονομαστικές τις υπερψηφίζω όλες. Bene, la ehm, Ωραία. Έκθεση τούν. Πρώτο μπλοκ, πρώτη ομάδα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, Έκθεση επιτροπή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η πρόταση επιτροπή. και σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Γκρέσ. Πρώτη ομάδα τροπολογιών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται πρόταση της Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Και με ονομαστική κλίση ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση τη Ρολιά. Τελευταία. 109 τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 13. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 13. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και με ονομαστική κλίση το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα γίνει μια διακοπή για την πανηγυρική συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε κατόπιν της ψηφοφορίας.